στα Ουγγρικά. Το επόμενο θέμα είναι η κοινή συζήτηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και επανεγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν έχουμε την έκθεση Reimer Böge, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση Βέλγιο, το Μέσκλο τη Ιφαντουργία και Ιρλανδία Ντέλ. Και μετά θα γίνει μια προφορική ερώτηση σχετικά με τι επαναγκαταστάσει επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν θα δώσω τον λόγο για τέσσερα λεπτά στον εισηγητή κύριο Μπέγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ως εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, υποβάλλω την ε, ε, έκθεση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής για δύο περιπτώσεις. Πρώτον, πάνω στις αιτήσει από